Ευχαριστώ πολύ ε, για τις ε, ουσίες προτεραιότητας. Δεν θα πω τίποτα γιατί νομίζω ότι το κλείσαμε το θέμα. Πέρα συζήτηση, πριν να περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να ενημερώσω ότι αρμόδιο στι αρχέ μα ενημερώνουν η κυρία Νόραμπερα, αντικαθίσταται από τον κύριο Μισελ Νταντέν, διότι η κυρία εξελέγει ε, ο κύριος Νταμιέ Ραβά και η κυρία Εστέρ ε, εξελέγησαν μέρη, μέλη της συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγραφος 2 που, αφορά την ε, εκλογή των μελών με καθολική ψηφοφορία. Αυτό υπάρχει ασύμβατο. Συνεπώ, οι θέσει είναι και να Η κυρία Ιζαμπέλ Μάξ εκλέγεται μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντικαθιστώντα τον κύριο Τωμά. Ο κύριο Ζαλουϊκοτινή εκλέγεται μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντικαθιστώντα την κυρία Εξτέλ Γκριγέ μέχρι τι 17 ε, ε, ε, Ο κύριο Νταντέν εκλέγεται μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντικαθιστώντα τον κύριο Ντανιέλα μέχρι από τι 17 Ιουνίου 2012. 12. Θα ήθελα να καλωσορίσω του νέου συναδέλφου και σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγραφό 2 του κανονισμού ε, θα πρέπει να γίνει ο έλεγχο των εξουσιών. Θα πρέπει να ελέγξουμε ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ο κύριο Γεντενή Περθιά ε, είναι μέλη του Κοινοβουλίου και έχουν ε, απολάμβουν των δικαιωμάτων του υπό τον όρο ότι θα δηλώσουν ότι δεν ασκούν κάποιοι. δεν, υπάρχει ασύλληβαστο. Περνάμε τώρα σε παρεμβάσεις του ενός λεπτού. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ζαμπόσκα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή για να θυμίσω ότι από χθες ξεκίνησε, ε, ετέθησαν ε, νέα ανώτατα σημεία. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς ε, μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Δεν θα ήταν δυνατόν